Przewodniczący! Uh, ah, αγαπητοί συναδελφοί, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Wznawiam sesję. Otwieram Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπη στις 17 Ιουνίου 2010. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 17 Ιουνίου και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Όχι, τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται. Θα ήθελα τώρα να σας ανακοινώσω πως σήμερα το πρωί επέστρεψα από επίσημη επίσκεψη στην Ρωσία. Η πρώτη επίσκεψη Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και 12 χρόνια. Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο Μετβέντεφ, τον Πρόεδρο της Δούμας Μπόρις Γκρίσλοφ, του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ρεσκέη Γκρίσλοφ και τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ενέργειας. Μιλήσαμε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-Ρωσία στο πλαίσιο της συνεργασίας για τον εξυγχρονισμό και την πιθανότητα νέας συμφωνίας ε, διμερούς. Ε, συζητήσαμε και άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης συναντήθηκα με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας ε, των πολιτών, μεταξύ των οποίων και της οργάνωσης Memorial που έλαβε το βραβείο Ζαχάροφ το 2009 κατά τη διάρκεια της παραμονής μου κλιμακώθηκε η διαφωνία με τη Λευκορωσία για το φυσικό αέριο. Διαβίβασα την ανησυχία μας στις ρωσικές αρχές και ζήτησα από τα δύο μέρη να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για την παράδοση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης σημείωσα πως ε, θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές ρήτρες στις συμβάσεις μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας που θα εγγυώνται την παροχή αερίου στην Ένωση. Η, παρο... η εγγύηση αυτή είναι το σημαντικότερο για εμάς. Επίσης, Κομισιόν και Συμβούλιο εξετάζουν το ζήτημα. Ίσως λοιπόν οι εκπρόσωποι θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αλλάζει, βρίσκεται εν εξελίξη. Κάθε ώρα έχουμε νέες πληροφορίες σε σχέση με αυτή την ε, διαφωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας βρίσκονται στα θεωρία. Τους καλωσορίζω ιδιαίτερα τον ε, κύριο Κεμάλ Αζίζ Σταμβουλέλ. Delegacja Indonezji w parlamencie η Ινδονησιακή Αντιπροσωπεία φιλοξενείται επ' ευκαιρία της ε, συνεδρίασης της διακοινοβουλευτικής ε, διάσκεψης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδονησίας. Ξέρετε πως πρόκειται για μια αναψώμενη οικονομία που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ΑΖΙΑΝ, την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πρόκειται για την πρώτη χώρα με την οποία υπογράψαμε το 2009 συμφωνία σύνδεσης και συνεργασίας και με μεγάλη ευχαρίστηση καλωσορίζω εδώ πέρα τους Ινδονήσιους βουλευτές. Επόμενο θέμα, προς ενημέρωση. Ο κύριος Μάικ Νάτρας έφυγε από το κόμμα της Ευρώπης για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία και από τις 23 Ιουνίου 2010 θα λογίζεται με τους μη εγγεγραμμένους. Επίσης οι αρμόδιες αρχές ε, της Ολλανδίας με πληροφόρησαν πως ο Λουίς Μπόντες αντικαταστάθηκε από τον Λούκας Χάρτονγκ και η κυρία Ζανίν Χενής Πλάσχερτ από τον κύριο Γιάν Μιούλτερ από τις 22 Ιουνίου 2010. Δηλαδή από χτες. Καλώς ορίζω τους ε, νέους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού μέχρι να επαληθευτούν ε, οι εντολές τους ο ε, κύριος ε, Λούκας Χάρτον και Γιάν Μίλντερ θα συμμετέχουν έχοντας ε, επίσης δηλώσει πως δεν έχουν κάποια, κάποιο άλλο αξίωμα που είναι ασυμβίβαστο με αυτό του Ευρωβουλευτή. γραμματεία των μη εγγεγραμμένων μου ανέφερε τις εξής ε, υποψηφιότητες για τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες. Για την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ο Λούκας Χάρτονγκ στη θέση του Ντάνιελ Φαντερστέπ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 της ε, σεξουαλικής παρενόχλησης έχει υπογραφεί αυτή η δήλωση οπότε συγχαίρω τους ε, συναδέλφους οπότε σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα δημοσιευτούν στα κείμενα τα οποία φτύθηκαν σε αυτή τη σύνοδο μαζί με τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2010. Καλωσορίζω λοιπόν τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας καλωσορίζω κύριε. Πριν περάσουμε στην ε, συζήτηση θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χερμάν Φαναρομπό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από όταν έγινα πρόεδρος, η οποία δεν είχε ως αντικείμενο κατεπήγοντα γεγονότα.